Το κείμενο αυτό θα ψηφιστεί αύριο. Μία ανακοίνωση. Βάσει του άρθρου 2.16 παράγραφος 4 του κανονισμού σας πληροφορώ ότι δεν έχω κανένα αίτημα για ψηφοφορία ε, της ε, ε, τροποποίησης η οποία, και της διόρθωσης η οποία έλαβε χώρα χθες, επομένως θεωρείται εγκεκριμένη.